Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την τιμή την δόκτωρα Αμάλα Αλκουμπάζη να συναντήσω, είχα την τιμή να τη συναντήσω. Είναι πρόεδρος του Κοινοβουλίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είναι προσκεκλημένη μας σήμερα και θέλω να την ευχαριστήσω, κυρία συνάδελφε. Ως πρόεδρος ενός Κοινοβουλίου μιας ε, μουσουλμανικής χώρας επιτύχατε να υπάρξει σαφής καταδίκη και καταθέσατε Στέφανο στο σημείο αυτής της αιματηρής επίθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι και σας καλωσορίζω. Πρώτα απ' όλα διαδικαστικά έχει ζητήσει ο κύριος Βέμπερ. Για διαδικαστικό ο κύριος Βέμπερ έχει ζητήσει το λόγο. Αναφέρομαι στο άρθρο 186 και το 11.2 του κανονισμού. Να υπενθυμίσω, προχθές μπροστά στην αίθουσα του Κοινοβουλίου έγινε ενός λεπτού σιγή και μία ε, σύντομη τελετή εις ανάμνηση των θυμάτων της τρομοκρατίας με πρωτοβουλία της Τερέζα Χιμένεθ από την πολιτική μας ομάδα. Και ο λόγος ε, για αυτήν την τελετή ήταν ότι σε μια συνεδρίαση της Γκουε παρευρέθηκε ο κύριος Οτέγγι, πρώην τρομοκράτης της ΕΤΑ. Είχε προσκληθεί. Είναι καταδικασμένος τρομοκράτης. Συμμετείχε στην συνεδρίαση της Γκουε και πήρε το λόγο για να συζητήσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΕΛΚ ζητάει να εξεταστεί αυτό το θέμα από την ε, πλευρά μας η ενόψη της μνήμης των θυμάτων είναι πρόκληση πρώην τρομοκράτες να παίρνουν το λόγο και να προσκαλούνται εδώ στο Κοινοβούλιο για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω επειδή ε, υπήρξαν τρομοκρατικές επιθέσεις πριν από λίγες μέρες ε, μπροστά στην πόρτα μας δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά τέτοια πράγματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαίνει δημοκρατία, ειρήνη, ελευθερία και πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι κατά της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Βέμπα. Ευχαριστώ κύριε Βέμπερ. Θα λάβω υπόψη αυτά που είπατε. Αναφερθήκατε στο 186 παράγραφος 2 ως αίτιο και πρέπει να το δεχτώ. Όμως πρέπει παράλληλα να σας πω ότι αγαπητοί συνάδελφοι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τώρα συζήτηση για ένα απλό λόγο γιατί πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία της Ολομέλειας ε, καταλαβαίνω έχω πολλές ε, επιστολές λάβει αλλά προσκλήσεις από ομάδες ή από βουλευτές ε, σε άτομα που άρα λαμβάνουν την δυνατότητα ε, να παρευρεθούν εδώ δεν είναι δική μου αρμοδιότητα ούτε κανός οργάνου εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί ε, λόγοι ποινικού περιεχομένου που μας αναφέρουν οι βουλευτές. Έχω κατανόηση για τα συναισθήματα αλλά κατά αυτής της ατομικής πρόκλησης δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι ένα θέμα πολιτικής αποτίμησης των μεμονωμένων βουλευτών ή των πολιτικών ομάδων εάν θα πρέπει να προσκαλούν ή όχι τέτοια άτομα. Ε, θα σας παρακαλούσα να ε, συζητηθεί το θέμα αυτό στη διάσκεψη των Προέδρων ή στο Προεδρείο στο οποίο θα αποστείλω το θέμα αυτό. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τσίμερ γιατί αναφέρθηκε η ομάδα της αλλά δεν θα δώσω σε κανένα άλλο το λόγο γι' αυτό γιατί δεν θέλω να ξεκινήσει συζήτηση γι' αυτό. Παρακαλώ κυρία Τσίμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω συζήτηση γι' αυτό, να διευκρινίσω τα εξή δύο. Πρώτον, είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τελεία. Αλλά πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άτομα τα οποία έχουν ε, εκφραστεί υπέρ μια διαδικασίας ειρήνευσης και παίζουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, αυτά τα άτομα θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στη δημοκρατική συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι Χιμένεθ. Αγαπητοί συνάδελφοι Χιμένεθ. Έχουμε κατανόηση για την κατάστασή σας και για την ε, τα συναισθήματά σας, αλλά επιμένω, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό τα αρμόδια όργανα και δεν θα δώσω σε κανέναν άλλο το λόγο από αυτού. Τα πρακτικά και τα εγκριθέντα κείμενα της συνεδρίας 14, Απριλίου είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά της συνεδρίασης της 14 η Απριλίου. Γι' αυτό συζητάμε. Όχι, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Τα πρακτικά